Good Καλημέρα, φίλοι μου. Θα ξεκινήσουμε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα με το πρόγραμμα. Ε, ξεκινήσουμε αμέσω. Θα έχουμε όλες τις γλώσσες, εκτός από τα τα Μαλτεζικά, τα Κροατικά και τα Γελικά. Επίσης, να ανακοινώσω ότι έχουμε και μια ομάδα 16 επισκεπτών που βρίσκονται εδώ ή θα έρθουν πολύ σύντομα και που έχει προσκαλέσει η κυρία Μωράν Σαρτιέ. Θα έρθουν εδώ για το πρώτο μισάωρο της συνεδρίασής μας και έχουμε και μια ομάδα 20 επισκεπτών που έχει προσκαλέσει η κυρία Σάντερ οι οποίοι επίσης θα έρθουν στις 9 και το απόγευμα θα έχουμε νέα νέους που θα παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Του έχει προσκαλέσει ο κύριος Λεϊαρίκ. Και θα έρθουν κανονικά στις 3.30. Ωραία. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ενημέρωση για την αποστολή της Επιτροπής μας στην, στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας στη Γενέβη, στον ILO. Ίσως η Γιούτα Στάινρουκ. Α, όχι, το αναβάλλουμε το σημείο αυτό. Γιατί όπως βλέπετε η επικεφαλής αντιπροσωπείας δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής θα οργανώσει ένα κοκτέιλ στις 13 στις 7 Δεκεμβρίου στον τρίτο όροφο του κτηρίου Γιάν στις 6.30 το απόγευμα. Και είναι προσκεκλημένοι όλοι οι εκπρόσωποι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από κυβερνητικές οργανώσεις και άλλοι. Ξεκινάμε λοιπόν με το σημείο 3. Ενημέρωση για τον Γιούρες. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φορέων Απασχόλησης. Όπως ξέρετε, ο κύριος Μπέκερ είναι ο εισηγητής, ο οποίος πέτυχε πολύ θετικά αποτελέσματα. Σας δίνω λοιπόν το λόγο για να μας παρουσιάσετε σύντομα το θέμα. Ε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω με έναν ε, τρόπο ε, με τον οποίο δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα στο παρελθόν να το κάνω. Ε, στο παρελθόν λοιπόν δεν βίωσα μια τόσο καλή συνεργασία και ήταν μια πάρα πολύ καλή ημέρα για την Επιτροπή Αποσχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να το πω εξ αρχής η πρωτοβουλία της Επιτροπής ε, για τη δημιουργία μιας νέας πλατφόρμας για το IRES ε, πάνω στο οποίο εργαστήκαμε. Ο στόχο, η στόχη ήταν κοινή να ε, ανυψώσουμε σε ένα νέο επίπεδο την πλατφόρμα ε, και ε, οι προτάσεις ε, της Κομισιόν τις οποίες αποφασίσαμε εμείς εδώ στο, στην Επιτροπή υποστηρίστηκαν ιδιαίτερως και θα ήθελα γι' αυτό να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι εργαστήθηκαν πάνω σε αυτό ιδιαιτέρως τον σκιώδη γνωμοδότη και, τον, και όσους έδωσαν συμβουλές οι οποίοι σε ένα πλαίσιο συνεργασίας κατέστησαν δυνατό αυτό, ούτω ώστε εμεί μαζί με το Συμβούλιο και την υποστήριξη ε, της Κομισιόν να μπορέσουμε να έχουμε ε, ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Τα βασικά στοιχεία λοιπόν από τη δική μας ε, πλευρά μπορούμε να τα περιγράψουμε με το ότι επιθυμούμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη, να ενισχύσουμε την κινητικότητα ούτως ώστε να υπάρξει, ώστε να μπορέσουμε να πολεμήσουμε και την ανεργία σε συγκεκριμένε περιοχές. Τα βασικά σημεία από την πλευρά ε, της Επιτροπής ε, μπόρεσα να τα παρουσιάσω ήταν ο ρόλος ε, των κοινωνικών εταίρων οι οποίοι έχουν επιδείξει μια ιδιαίτερη σημασία και η ποιότητα των συνεισφορών τους ήταν πάντοτε ε, άριστη προς την αγορά εργασία. Ένα άλλο σημαντικό σημείο το οποίο επεξεργαστήκαμε ήταν η δομή να ε, δημιουργηθεί έτσι ούτω ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε ε, επαγγελματικές ποιότητες προς τα Ευρωπαϊκά Γραφεία Συντονισμού, προς τα Εθνικά Γραφεία Συντονισμού μαζί με τους ε, εταίρους ε, και τα μέλη καθώς επίσης και με τους ε, συνεργάτες δηλαδή το προσωπικό το οποίο μπορεί να είναι σίγουρο ότι θα έχει μια άριστη κατάρτιση δώσαμε ιδιαίτερη βάση λοιπόν στην ποιότητα των διασυνοριακών συνεργασιών, των μεγάλων συνεργασιών που έχουν δημιουργηθεί και εδώ πέρα έχουν ε, μια ιδιαίτερη βάση και με τα χαράς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησε την ευθύνη του με το ότι έδωσε στην Επιτροπή Αποσχόλησης ε, κάθε βοήθεια ούτως ώστε αυτό το άριστο ε, έργο και πρόγραμμα της Κομισιόν να μπορέσει να υποστηριχθεί από τα κράτη-μέλη μετασιγουριάς ε, θα είναι παρο... νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσω συγκεκριμένα άτομα τον ε, ε, πρόεδρό μας των τριμερών διαλόγων που συνεισέφερε ιδιαιτέρως σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω Ιδιαίτερα πρέπει να ευχαριστήσω και την ε, Βάρβαρα από την Γραμματεία, η οποία έκανε πολύ καλό έργο. Θα μπορούσα ε, να ε, ήμουν και πιο σύντομος. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τις νομικές υπηρεσίες με τον Μάριο και θα ήθελα να αναφέρω και την Ελίνα η οποία παρεπιπτόντως σήμερα έχει τα γενέθλιά της και δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι ε, σύμπτωση ότι το καλύπτει σήμερα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι για την ποιότητα της εργασίας αυτής ιδιαίτερο ρόλο έπεσε, έπαιξε η συνεργασία. Ε, θα ήθελα επίσης να αναφέρω τον ε, Σίμον, την Γιάννη Τσιλάντσκα, την Πορίνα, την Ματίνα Κλάπαγιόβα, Γκουε Παλώμα, Αντνέτε Μπόγκα, καθώς επίσης και από τους πράσινους Σλέτσεβιτς, ε, Λαουρα Γκέα. Εσείς όλοι έχετε συνεισφέρει πάρα πολλά σε αυτό και αυτό φαίνεται και, από, και σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε και την ποιότητα των εταίρων όπως είναι ο Εμμανουέλ Ματιό και ο Σλίμ από το Συμβούλιο. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα. Εδώ έχω την γραβάτα από το Λουξεμβούργο, από την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Ε, είχαμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και τέλος αλλά όχι έσχοτο η ε, Κομισιόν ε, Σάκη Μορέν και την ομάδα της ε, και εδώ θα σταματήσω εδώ και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ και ελπίζω να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτή την επιτυχία σας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέκερ. Πολύ ενδιαφέρον το ταξίδι που μας κάνατε. Το αποτέλεσμα που πετύχατε θα το ψηφίσουμε σύντομα. Επιτυχία όμως σημειώσαμε και στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πυρίνσκι που θα μας παρουσιάσει την ανακεφαλαίωση των όσων έγιναν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά επιβεβαιώνω όσα είπατε. πετύχαμε να έχουμε συμφωνία για τη δημιουργία πλατφόρμας για να αντιμετωπίσουμε και να αποτρέψουμε την αδίλωτη εργασία. Ξεκίνησαν από τον Απρίλιο σχετικές συζητήσεις όταν υπέβαλε την νομοθετική της πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τον Μάιο εμείς ψηφίσαμε τη θέση μας. Μετά ξεκίνησαν οι διπραγματεύσει με επικεφαλή σα κυρία Πρόεδρε και ο τριμερής διάλογος έγινε σε πρώτη φάση με τη Λετωνική και μετά με τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Στις 11 Νοεμβρίου μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο και στις 20 του ίδιου μήνα ενημερωθήκαμε ότι το Κορεπέρ δέχτηκε όσα πετύχαμε και συμφωνήσαμε. Δεν θα απαριθμίσω όλες τις λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν, κάνουν ξεχωριστή αυτή την πλατφόρμα αλλά θέλω να επισημάνω το τι θέλουμε να μας προσφέρει αυτή η πλατφόρμα. Συγκεκριμένα λοιπόν θέλουμε να μας προσφέρει συμπεράσματα. Συμπεράσματα για το πώς να αποτρέψουμε και να καταπολεμήσουμε την αδηλωτή εργασία, αλλά ταυτόχρονα πώς να τη μετατρέψουμε σε εργασία δηλωμένη, νόμιμη. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτό το στοιχείο, τα συμπεράσματα, τα πορίσματα, γιατί αυτή είναι η επικοδομητική ε, λύση που πετύχαμε μεταξύ δύο διαφορετικών σημείων αφετηρίας. Όπως τα γνωρίζετε και εσείς και οι συνάδελφοι, υπήρχαν διασμοί σε πολλά κατημέλη και σε πολλέ πολιτικέ ομάδε, εάν υπάρχει πραγματικά ανάγκη για τέτοια πλατφόρμα. Διότι αυτό θα ήταν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Επίσης, κάποιοι αισθάνονταν ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να έχει και ρυθμιστική λειτουργία. Νομίζω το αποτέλεσμα που πετύχαμε είναι πολύ λειτουργικό, πολύ εύστοχο. Υπάρχει εκπροσώπηση από τα κράτη-μέλη με υπευθυνότητα στα ανώτερα κλιμάκια εκπροσώπησης. Επίσης τέσσερις κοινωνικοί εταίροι με ισότιμη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις μας ε, οδήγησαν στο σωστό αποτέλεσμα και υπάρχει και ένα ευρύ φάσμα παρατηρητών που θα μπορούν να συμμετέχουν στην πλατφόρμα. Κατά αυτόν τον τρόπο Νομίζω ότι καλύψαμε τις ανησυχίες και των συναδέλφων με τους οποίους είχαμε συζητήσει και εδώ στην Επιτροπή και των κρατών μελών που φοβούνταν ότι μπορεί να υπήρξε παραβίαση ή παρέμβαση στις εθνικές τους αρμοδιότητες. Ταυτόχρονα η μορφή αυτή που συμφωνήσαμε μπορεί να επιλύσει πολύ γρήγορα, κατεπήγοντα και καυτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αδήλωτη εργασία. Κοιτάζοντα αρχικά του ορισμού τη αδήλωτη εργασία, διότι ο κλασικό ορισμό από τα τέλη τη δεκαετία του 1990 δεν είναι πλέον επίκαιρο, ούτε αρκετά συγκεκριμένο και επίσης τις δράσεις που θα αναλάβει η πλατφόρμα και που συζητούνται. Υπάρχει μια ποικιλία από αυτές για την ανταλλαγή πληροφοριών, για τις βέλτιστες πρακτικές, για να ανταλλάσσονται ιδέες και προσεγγίσεις και πώς κατά τον καλύτερο τρόπο μπορεί να αντιμετωπίζονται διάφορες μορφές αδήλωτης εργασίας. Εδώ, Πρόεδρε, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μπέκερ, εκφράζοντας και τη θερμή ευγνωμοσύνη προς τους συναδέλφους και την διαπραγματευτική ομάδα από όλες τις πολιτικές ομάδες. Η συμμετοχή τους ήταν πολύ ενεργή και των ίδιων και των συνεργατών τους. Θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματεία. Δίπλα σας κάθεται ο Καλή Μόιρα. Μας βοήθησε πάρα πολύ με, πολύ, τις πολύ ακριβείς περιλήψεις και ανακεφαλαιώσεις της στην όλη διαδικασία. Και ο Γιάνν Τρόμς από την Γραμματεία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ήταν πολύτιμη βοήθεια και η νομική υπηρεσία και όλοι οι συνεργάτες που ανέφερε και ο κ. Μπέκερ. Να αναφέρω ότι είχαμε και πολύ επικοδομητική συνεργασία με την Προεδρία του Λουξεμβούργου. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι η Προεδρία αυτή το κοινωνικό θεματολόγιο το έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα και με τους εκπροσώπους της Προεδρίας από τον τριμερή διάλογο είχαμε πραγματικά ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας για να βρούμε τις κατάλληλες συμβαστικές λύσεις. Γι' αυτό, Πρόεδρε, Πιστεύω ότι η τελική συμφωνία που πετύχαμε και απαραίτητη ήταν και θα μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά και θα είναι και μια σοβαρή συνεισφορά στην αντιμετώπιση αυτών των πολύ μεγάλων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αγορά εργασία στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το συμπερασμά μου. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. you, Ευχαριστώ κύριε ε, Πινιένσκι και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ερωτήσεις ε, προς τους ομιλητές τότε υπάρχει δυνατότητα ε, να θέσετε τώρα τις ερωτήσεις. Έχουμε τέσσερα λεπτά πριν ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Yes, Laura Agia. Ναι, η Λάουρα Άτζια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπέκερ, διότι ήταν εξαιρετική η δουλειά του και έδωσε σε όλους τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Όταν θα πάρει την τελική του μορφή το έγγραφό μας, Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το προβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Να το γνωστοποιήσουμε σε όσους θα χρειαστεί να το αξιοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή το Γιούρες δεν έχει αρκετή προβολή και δεν, έχει αρκετή, δεν είναι αρκετά γνωστό. Χθε μιλούσαμε με φοιτητές του Πανεπιστημίου της Περούτζα και του ρωτούσα αν γνωρίζουν αυτή την πλατφόρμα δυστυχώς δεν την γνωρίζανε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, τι μπορούμε να κάνουμε για να διαδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτήν την πλατφόρμα. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να, να φανεί πολύτιμο, αλλά εάν δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, αυτή η πολύ ωραία προσπάθεια δεν θα έχει την επιτυχία που θέλουμε. We'll have to vote in minutes. Θα ψηφίσουμε σε δύο λεπτά, αλλά ένα πολύ σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Απλώς να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Μπέκερ, κύριο εκείνον, για τη δουλειά του. Διότι διοργάνωσε πολύ καλά ό,τι χρειάστηκε να κάνουμε από κοινού για το δίκτυο Γιούρες. Ευχαριστώ και τους εμπειρογνώμονες, μάλλον τους συμμετέχοντες σε όλη την ομάδα, διότι βλέπω εδώ ότι όταν υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιο θέμα μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα και τους στόχους μας. Πολύ γρήγορα, κυρία Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω εσάς και όλους τους συναδέλφους που μας αποκλείσατε από τα δύο αυτά θέματα, παρόλο που την ομάδα μας την έχουμε συστήσει εδώ και έξι μήνες τουλάχιστον. Well, you could have, appointed Mr. Martin Έχετε ε, ένα δίκαιο κύριε Μαρτάν. Ε, δεν διορίσατε κάποιον και γι' αυτό το λόγο δεν λάβατε τις πληροφορίες. Δεν είναι έτσι στις συνεδρίες των συντονιστών. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό. Στην ίδια σειρά έχει το λόγο η συνάδελφος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, επειδή αντικαταστώ τη συνάδελφο σήμερα, Σα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Βάσει των πληροφοριών που έχω εδώ, ο προπολογισμό, το κονδύλι, προβλέπει 2,1 εκατομμύρια και 224.000 για τα TND. Έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένε λεπτομέρειε για το τι θα επιτραπεί και θα γίνει και έλεγχος λογιστικός για να είμαστε βέβαιοι ότι τα κονδύλια αυτά δαπανήθηκαν σωστά και όπως δει. Ε, θα έλεγα και η δική μου συμβουλή θα ήταν να μιλήσετε με το σχέδιο συγκεκριτή τη ομάδα σας για να έχετε όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες. Ο κύριος Κάζα. Just a small point, Madam Chairman. Κάτι που θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση, όμως θα πρέπει να δείξουμε μια, ένα σεβασμό στην Προεδρία και υπό καμία ε, κατάσταση δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ψέμα, ε, ίσως μια παρανόηση, όμως θα πρέπει να είμαστε γενικά κάπως προσεκτικοί το πώς μιλάμε σε εσά και οποιοδήποτε άλλο Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κάζα. Θα ψηφίσουμε τώρα. Ελπίζω να έχετε τις κάρτες σας. Mm. Okay, you seem to be ready. Then Φαίνεται να είστε έτοιμοι. Έχετε τις κάρτες σας για να ψηφίσετε. Οπότε θα ψηφίσουμε το συμβαστικό κείμενο που πέρασε και από το Κορεπέρ για πρώτες απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την ενίσχυση της αποτροπής και καταπολέμησης της αδίκοτης εργασίας. Ξεκινά η ψηφοφορία. Ένας υπεράριθμος στο ΕΛΚ. Στο ΕΛΚ υπάρχει ένας παραπάνω που ψηφίζει. «45 υπέρ, δύο κατά». Τελική ψηφοφορία για το Γιούρες. Υπηρεσίες απασχόλησης. Απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Σαραντατέσσερις υπέρ και Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Χειροκροτήματα. Χειροκροτήστε τον κύριο Πυρίνσκι παρακαλώ. Okay, then we proceed with the... Και τώρα, κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, Προγραμματισμό κομπιούτερ από τη Φινλανδία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 42 προ 5. Επόμενο σημείο, δεύτερο η PWA International της Ιρλανδίας άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 42 προς 5. Σημείο 6 πολιτικές καταπολέμησης της ενεργειάς των νέων, πολιτικές ανάπτυξης δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της ενεργειάς των νέων. Συμβιβαστική ή ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Κατά. Εβδομήντα δύο. Παράγραφος 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές αποδεκτό. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές δεκτό. Σελίδα 5 18 υπέρ κατά αποχές δεκτό 28 υπέρ κατά αποχές δεκτό 19 υπέρ κατά αποχές 88 παραγραφός 3 υπέρ κατά αποχές δεκτό παραγραφός 3 υπέρ κατά αποχές απορρέπτεται παραγραφός 3 τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβιβασμός 98 και 99 μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παραγραφός 4 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Παράγραφος 4 101 υπέρ κατά αποχές δεκτό 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 και 4 παράγραφος 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά έλεγχος 106 πέρας 21 προς 24 απορρίπτεται. 30 της Επιτροπής Κούλτ για την παράγραφο 5, νέα εκδοχή υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κούλτ 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 107, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 15 σελίδα 8, όχι, 120 παράγραφος 6α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 Παράγραφος 6α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική J. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική και η κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138. Παράγραφος 8, σελίδα 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κουλτ 34, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κουλ 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 και 147 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Συμμεβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμμεβαστική T σελίδα 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 2 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική. 159. πενήντα Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 161 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 170 και 171 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Κουλτ 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ε, 172. 27 προς 26 εγκρίνεται. Συμβαστική ο, όμικρον. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κουλτ 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. ...236 υπέρ, κατά... ...236... ...α, η 33 εννοείται... ...η 33 καταπίπτει... ...οπότε ψηφίζουμε την 236... ...και πάλι ποιοι είναι υπέρ... ...ευχαριστώ, κατά εγκρίνεται. 183. 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Κουρτ 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κουλτ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουρτ 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Κουλτ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205 και 206 μαζί υπέρ κατά 207 μαζί με την τροπολογία και αυτή υπέρ κατά αποχές 207 λήξη της ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι 29 κατά, 25 υπέρ. Απορρίπτεται λοιπόν, οπότε περνάμε στο 208 υπέρ κατά, αποχές, ε, δεκτό. Καλτ ε, υπέρ κατά, δεκτό. 218 υπέρ, κατά, αποχές δεκτό. 219 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Υπέρ, κατά. Συμβιβασμός U, υπέρ, κατά, δεκτό. 228 υπέρ κατά αποχέστε δεκτό συμβιβασμός σταυλιού υπέρ κατά ε, αποχέστε δεκτό τροπολογία δεκτό 234 υπέρ κατά συμβιβαστικό υπέρ κατά αποχές συμβαστική υπέρ κατά συμβαστική on page 24. Yes, 24. Those in favor. Υπέρ κατά αποχές δεκτό 253 υπέρ κατά συμβαστική 254 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 256 υπέρ κατά απορρίπτεται 257 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 257 Συμβαστική 259 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Q ...261 στη σελίδα 26. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 260 όχι, πάμε κατευθείαν στις αναφορέ. Ε, αναφορές. Ε, αιτιολογική αναφορά 1 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Το 2 και 3 μαζί, αυτή υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 4 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 5 και 6, 8 και 9, υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, ε, Recital 11 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 18 υπέρ κατά εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται υπέρ κατά εγκρίνεται 23 υπέρ κατά εγκρίνεται 24 υπέρ κατά απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 26 υπέρ κατά απορρίπτεται Το 27 απορρίφθηκε, οπότε πάμε στη συμβαστική B, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 30, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγξτε την τροπολογία 39 λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται για μία ψήφο. Περνάμε στη συμβαστική D. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στο 46 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, απορρίπτεται 50 υπέρ κατά εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά απορρίπτεται 53 υπέρ κατά εγκρίνεται 54 υπέρ κατά εγκρίνεται και τώρα θα ψηφίσουμε ε, για το σχέδιο της αναφοράς το οποίο τροπολογήθηκε. Ψηφίσατε. Λήξη ψηφοφορίας. 49 υπέρ. Μία κατά. Congratulations to You did a good work. Συγχαρητήρια, κάνατε πολύ καλή δουλειά και το αποτέλεσμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην τελική αναφορά ε, η οποία, την οποία ετήθηκε το 1 τρίτο των ε, μελών που παρευρίσκονταν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Συμφωνείτε λοιπόν σε αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δεν υπάρχει σλοβακική διερμηνία διότι ο διερμηνέας έχει αρουστήσει. Οπότε θα πρέπει να ακούτε ε, άλλες γλώσσες. Ah, okay. Uh, then we proceed uh, to... Um, Uh, the draft opinion, uh, my... Περνάμε τώρα στο σχέδιο έκθεσης της κυρίας Γκουνσάλες Πένιας και ψηφίζουμε. Συμβιβαστική Α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική B υπέρ, κατά, αποχές. Μάλλον πρέπει να ελέγξουμε. Τώρα σηκώνατε τα χέρια σας. Οπότε δεν θα χρειαστεί να ψηφίσουμε. Μάλιστα, εγκρίνεται. Τροπολογία, όχι, συμβαστική C υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Πέρας. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 να κάνουμε και έλεγχο. And the vote is now... Και έτσι πέρασε ψηφοφορία. Όχι, Πώ είπατε. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Γέλια στην αίθουσα. E. Συμβαστική C, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές ε, γκρίνεται. Η H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική ΑΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αν θέλετε την 102 να την ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. 102 ελέγχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 103 παρακαλώ. Πέρας. 103. Βλέπετε 26-26. Τροπολογία 104 και 105 μαζί. Υπέρ των δύο. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική J, λατινικό υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική K, λατινικό υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε για να δούμε Πέρασες της ψηφοφορίας εγκρίνεται εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την 121, δεν βλέπω καθαρά το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Ψηφίζουμε, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 25-22. Το QA λατινικό υπέρ κατά η συμβαστική αυτή αποχές εγκρίνεται η συμβαστική MA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η L λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 132 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 132 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Από το ΕΛΚ ένας έχει ψηφίσει παραπανήσιος. Ακόμα ένας παραπάνω είναι. Απορρίπτεται. 23-27 το αποτέλεσμα. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική CA λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 138 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική, α, να ελέγξουμε, κάποιος ζητάει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 138. Ψηφίζουμε παρακαλώ, 138. Πέρας. εγκρίνεται 26-24. Συμβαστική εν λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...151 τροπολογία υπέρ... ...κατά... ...αποχές απορρίπτεται... ...154 υπέρ... ...κατά... ...αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε την 154 παρακαλώ. 154 ψηφίζουμε, πέρας. Εγκρίνεται 29-17. 156 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέξουμε την 157 παρακαλώ ψηφίζουμε λοιπόν 157 πέρας Δεν, δεν, δεν είδα τους αριθμούς εδώ πέρα. Το αποτέλεσμα εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 158. Ψηφίζουμε 158. Πέρας. Εξακολουθεί να ψηφίζει ένας παραπάνω από πλευράς ΕΛΚ. Για να το δούμε. Εγκρίνεται. 30-21. 159 υπέρ. 159 είπαμε υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ο λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η εκατόν, μισό λεπτό, μισό λεπτό η εβδομήντα, ναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, πι λατινικό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 177 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 178 179, 180 και 181 υπέρ αυτών των τεσσάρων υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, compromise Q. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 185, ξεκίνησε η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας για την 185 και εγκρίνεται. Τροπολογία 186 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 187 υπέρ, κατά, δεκτή. 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε ξεκίνησε η ψηφοφορία για την τροπολογία 190 λήξη ψηφοφορίας και εγκρίνεται για μία ψήφο Συμβιβαστική HA υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 194 Πάμε στην 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Και περνάμε τώρα στην ε, τροπολογία 1, υπέρ κατά εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Και τώρα στην συμβιβαστική R, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ κατά εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική S υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε τη 15, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για την τροπολογία 15. Εντάξει, έληξε, οπότε υιοθετήθηκε. Η ψήφο σα δεν μπορούσε να κάνει τη διαφορά σε αυτή την ψηφοφορία. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 18. Άρχεται η ψηφοφορία, έληξε για την τροπολογία 18 και εγκρίνεται για δύο ψήφους. Στην 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ όχι 24 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε την 24 Αρχιετή ψηφοφορία λήξη και εγκρίνεται συγγνώμη δεν το είδα 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία λήξη εγκρίνεται για δύο ψήφου και περνάμε στη συμβαστική τι, υπέρ κατά από ποια εγκρίνεται τροπολογία 36 υπέρ κατά ποια εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές θα έλεγα απορρίπτεται αλλά ας το ελέγξουμε ελέγχουμε την τροπολογία 40 έναρξη της ψηφορίας λήξη εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 ναι απορρίφθηκε 40, ε, ε, συμβιβαστική U υπέρ κατά εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε, 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα το ελέγξουμε Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. «58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, ελέγχουμε την 58, ε, έναρξη της ψηφοφορίας, Ελέγχουμε την 58. Λήξη της ψηφοφορίας. Και απορρίφθηκε. Τροπολογία 59. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 63. Υπέρ,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 και τώρα θα ψηφίσουμε σχετικά με το σχέδιο γνώμης όπως τροπολογήθηκε και ξεκινάει η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 43 προς 6. Then we'll go to... Οπότε θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία για την ε, ΤΙΣΑ. Uh, uh, να σας πω κάτι πριν ε, ψηφίσουμε. Γνωρίζετε ότι ο εισηγητής κύριος Χέντελ, ε, όπως βλέπετε δεν μπορούσε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη συνάντηση και ψηφοφορία. Όμως θα ήθελα να τον ευχαριστήσω παρόλο που δεν ε, είναι ανάμεσά μας. Ήταν μια άκρως επικοδομητική ε, συζήτηση για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση και νομίζω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε ένα καλά ισορροπημένο αποτέλεσμα και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες που συνεργάστηκαν ε, για να εξευρεθεί ένα αποτέλεσμα. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι όλοι μαζί. Γι' αυτό σας ευχαριστώ όλους σας. Οπότε πάμε στην ψηφοφορία. Τοπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F. Υπέρ. Κατά. Αποχές και θα ελέγξουμε τη συμβιβαστική F. Έναρξη λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε για μία ψήφο. Συμβιβαστική C. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική A υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε τη 17. Έναρξη της ψηφοφορίας λήξη για την τροπολογία 17 και απορρίπτεται. Συμβιβαστική H υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική HA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική HP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική Ι e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται νομίζω όμως μπορούμε να το ελέγξουμε σχετικά με την τροπολογία 34 λήξη της ψηφοφορίας απορρίφθηκε κατά τέσσερις ψήφους συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές πρέπει να το ελέγξουμε την τροπολογία 47 λήξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 47 απορρίφθηκε με 22 ψήφους και 21 που απήχαν. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε την τροπολογία 32. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται κατά τρεις ε, ψήφους και πάμε στη 48 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να την ελέγξουμε έναρξη της ψηφοφορίας λήξη εγκρίνεται με μία ψήφο. Τροπολογία 50 υπέρ για την τροπολογία 50 κατά αποχές απορρίπτεται τροπολ... συμβιβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική KA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές Ας την ελέγξουμε αυτήν. Συμβιβαστική L. λήξη της ψηφοφορίας για τη συμβιβαστική L παράγραφος 5 και εγκρίνεται Τροπολογία 66. Εφόσον η 65 ε, απορρίφθηκε, οπότε αποσύρθηκε, οπότε στην 66. Υπέρ, κατά, αποχές συγκρίνεται. Η 68 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την 68 έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε για δύο ψήφους. Τροπολογία 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ελέγχουμε την τροπολογία 79 έναρξη της ψηφοφορίας Ψήφισε και ο κύριος Μαν. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Η 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. δεν ψηφίζεται όπως συνήθως. Τροπολογία 83 υπέρ, κατά, αποχές. Πιστεύω ότι πρέπει να την ελέγξουμε την 83. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική ΟΟΥ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ελέγχουμε την τροπολογία 94 Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται με πέντε ψήφους. Συμβιβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική QA υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε τη συμβιβαστική QA ενέργεια της ψηφοφορίας. Λήξε. Εγκρίθηκε με μία ψήφο. Τροπολογία 97 υπέρ. Για την τροπολογία 97 θα κάνουμε δύο ε, ψηφοφορίες υπέρ ε, για το πρώτο κομμάτι κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο ε, κομμά, ε, κομμάτι υπογραμμίζει μέχρι κοινωνική εταίρη υπέρ κατά αποχές. Δεν μπορώ να δω, οπότε θα ψηφίσουμε για το δεύτερο κομμάτι, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. περίρο. Όμως εγκρίθηκε. Τροπολογία 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα η τελική ε, ψηφοφορία σχετικά με το ε, σχέδιο της ε, γνωμοδότησης με την τροπολογία. Λήξη της ψηφοφορίας. 38 υπέρ και 11 κατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάει ιδιαίτερως όταν είμαστε ενωμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Friends, we still have a... Έχουμε ακόμα μια συνάντηση, μια συνάντηση της Επιτροπής στην οποία θα προχωρήσουμε τώρα. Έχουμε αρκετά σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης έχουμε ε, την ε, ετήσια αναφορά ε, σχετικά με την εφαρμογή της συνοσιακής νομοθεσίας για την απασχόληση θέλουμε τώρα να ακούσουμε την συντάκτρια της γνωμοδότησης και θα δώσω τώρα το λόγο σε εσάς.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 Θα ήθελα να σας μιλήσω λοιπόν για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζει κάθε χρόνο μια τέτοια αναφορά. Τα κράτη-μέλη έχει νομοθεσίες που επιτρέπουν περισσότερες φορές το χρόνο να ελέγξουμε διάφορες ε, προόδους σχετικά με την ε, κοινωτική νομοθεσία σχετικά με τις εφαρμογές ε, των οδηγιών που έχουν καθυστερήσει οδηγούν σε ε, προβλήματα εάν, εάν εφαρμόσουμε τις ε, συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα ζητήματα τότε και οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν να υποφεληθούν από αυτό. Οπότε ε, παρατηρούνται οι σημαντικότερες ε, προόδοι ε, όταν αφορά το προηγούμενο χρόνο. Σχετικά με το 2014 είχαμε πάνω από 3.000 νέες διαμαρτυρίες στον τομέα της απασχόλησης και κοινωνικών ζητημάτων συνολικά 666 αφορούσαν την απασχόληση και οι περισσότερες αφορούσαν την κοινωνικότητα των εργαζομένων και ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Τώρα όσον αφορά την ίδια την αίτηση, θα ήθελα να σημειώσω ότι η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ελέγχει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ε, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κάτι ωφέλιμο για όλους μας. Το 2014 η Κομισιόν είχε τον μεγαλύτερο αριθμό ε, διαμαρτυριών ε, σχετικά με την απασχόληση. και η Επιτροπή αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι όσον αφορά την αξιολόγηση της νομοθεσίας ε, προσέξαν ιδιαιτέρως όταν αφορούσε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπρόσθετα το θέμα είναι η εφαρμογή της συγκεκριμένη νομοθεσίας και η βελτίωση ε, αυτού και εδώ μπορούμε να έχουμε διάφορα μέτρα όπως ετήσιες ε, ε, ενδείξεις, πίνακες αντιστοίχησης και είναι πάρα πολύ καλό εάν η Επιτροπή μαζί, μαζί, μαζί με τα κράτη-μέλη συνεργαστούν καλύτερα ούτως ώστε να επιταχύνουν την διόρθωση της νομοθεσίας. Επιπρόσθετα πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τις διαγνωστικές για ποιο λόγο έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα γίνει καλύτερα αν μπορέσουμε να εξετάσουμε για ποιο λόγο έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις διότι με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε και την ποιότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα λοιπόν οι ε, νομοθεσίες που δεν είναι ε, επίκαιρες θα πρέπει να ανανεωθούν ε, για παράδειγμα και και να εναρμονιστούν όλα αυτά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως το θέμα δεν είναι να έχουμε υπερβολική νομοθεσία, έχουμε διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια στα κράτη-μέλη και αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να υπάρξει μια παθητική αντίσταση από την πλευρά των κρατών μελών. Νομίζω ότι μια έγκαιρη ε, συνεργασία μεταξύ του ε, Κομισιών και των κρατών μελών θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος των ε, Σον Σάιμον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την πολύ χρήσιμη αυτή η γενική επισκόπηση. Νομίζω ότι το κείμενο που προτείνεται είναι καλό. Απλώς μερικά σύντομα σχόλια για ένα-δυο σημεία όπου μπορούσε να βελτιωθεί ενδεχομένως. Στους σοσιαλιστές και δημοκράτες θεωρούμε ότι ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερομένων πρέπει να αναφέρεται πιο έντονα στο κείμενο και με την παρακολούθηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποβολή εκθέσεων και την παρακολούθηση τη μεταφορά του κοινοτικού δικαίου από τα κρατη και Αυτά όλα πρέπει να είναι σαφή στο κείμενο. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κατά την εκπόνηση νέα νομοθεσία που θα αφορά τι μικρομεσαίε επιχειρήσει για περισσότερε 85% περισσότερε θέσει εργασία, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο του οικονομικού παράγοντε και τις, τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά και μακροπρόθεσμα τι μπορεί να γίνει. Πώ θα επηρεαστεί η αξία και τι κοινωνικά ωφέλη μπορεί να προσφέρει η νομοθεσία που θα προταθεί. Το κείμενο αναφέρει ότι το 2014 η Ένωση, μάλλον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έλαβε το μεγαλύτερο αριθμό προσφυγών, αλλά ταυτόχρονα να σημειώσουμε ότι στο τομέα τη απασχόληση των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής ένταξης δεν υπήρξαν καθόλου προσφυγές εκεί. Σχεδόν. Και τέλος, ίσως και το πλέον σημαντικό, πρέπει να τονίσουμε όπως ανέφερε και η συγγήτρια, τις συνέπειες της πραγματικής ε, παρακολούθησης και υλοποίησης και της έγκαιρης ε, μεταφοράς και της αντιμετωπίσης των ε, ελλείψεων. Δεν υπάρχει λόγος εκπόνησης νομοθεσίας, κανείς δεν κάνει τίποτα και δεν λειτουργούν τα πράγματα αυτά, όπως με την απόσπαση των εργαζομένων και τη σχετική οδηγία σουηδική λόγου χάρη παρέκκληση από την οδηγία αυτή. Όταν βρέθηκαν ελλείψεις και χάσματα θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν δράση με πολύ μεγαλύτερη πυγμή. Ιδάλλως δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπασί από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Συνάδελφοι, να ευχαριστήσω το, την εισηγητρία για την ε, δουλειά της στην έκθεση αυτή, τη γνωμοδότηση αυτή. Πολλές από τις δικές μας προτάσεις έχουν καλυφθεί. Θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια ότι αυξημένη επιρροή των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας θα ήταν ε, ωφέλιμη. Αν θέλουμε να αντικατοπτρίζει η κοινοτική νομοθεσία τις ε, τάσεις της πραγματικότητας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι συνθήκες επικρατούν σε επίπεδο κρατών μελών. Εάν αυτό δεν αντικατοπτρίζεται καλύτερα κατά τη ε, διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ιδίως κατά την υλοποίηση του ενωσιακού δικαίου. Οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές στηρίζουν τις πρωτοβουλίες για την καλύτερη νομοθεσία και την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σαφήνεια και λειτουργικότητα ε, για, ε, για την κοινωτική νομοθεσία. Ε, το θεματολόγιο της καλύτερης, της νομοθέτησης και η διαθεσμική συμφωνία είναι γαλέ ευκαιρίε για να μπορέσει πραγματικά η κοινοτική νομοθεσία να επιτυγχάνει το σκοπό που επιδιώκει. Το να έχουμε σαφή νομοθεσία θα αυξήσει το επίπεδο συμμόρφωση, την ταχεία μεταφορά και θα μειωθεί και το γραφειοκρατικό άχθο. Χαίρομαι ιδιαίτερω που βλέπω την εισηγήτρια να αναγνωρίζει ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να μην υπάρξει υπερβολικό άχθος από την κοινωτική νομοθεσία εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως σωστά εντοπίζει ε, είναι αυτές που δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας οι μικρομεσαίες. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι η αρχή του Think Small First, να σκεφτόμαστε πρώτα δηλαδή τους μικρούς, εφαρμόζεται και στην νομοθεσία μας, ιδίως προς τον Νότο κατά την άποψή μου. Η ομάδα μας Επίσης στηρίζει πλήρως τις πρόσφατες προτάσεις για μια ετήσια έκθεση για το γραφειοκρατικό άκθος όπου να δείχνει πού παρεμποδίζει η νομοθεσία μας την οικονομική ανάπτυξη. Και πάλι ευχαριστώ την εισηγήτριά μας για τη δουλειά της, νομίζω ότι η γνωμοδότηση είναι πολύ καλή και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Thank ε, Ευχαριστώ. Από τους φιλελευθέρους. Παρακαλώ. Κανείς από την Άλντερ. Πάμε στην ΚΟΕ. ΚΟΕ Η κυρία Λόπες Μπερνάγιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή για τη σωστή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης. Ε, είναι ένα σκληρό θέμα, αλλά είναι σημαντικό στο εργασιακό δίκαιο και για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτός ο ουδέτερος τόνος με εξέπληξε από πλευράς της συγγήτριας στο θέμα αυτό. Εμείς καταγγέλουμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν, αγνοούν τους νόμους ε, με το δικαίωμα ας πούμε μιας σε ένα χρόνο, ε, με συγγνώμη μια μέρα είτε τις διακοπές κλπ. Και στην Ισπανία υπάρχει μια καθυστερημένη, πανταργοπορημένη εφαρμογή αυτών των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια σκληρή πίεση λόγω της πολιτικής λιτότητας και επειδή παραβιάζονται οδηγίες για το χρόνο εργασίας, για μην ίση αντιμετώπιση ανάλογα με την κάθε κατηγορία εργαζομένων, με τις διακοπές κλπ. Και αυτό θα πρέπει να το πούμε κατά την απόψή μου στην έκθεση μέσα. Η μία εφαρμογή αυτών των νόμων είναι κάτι, μια επίθεση κατά των γενικών κατα των κοινωνικών υποθεσεων και στον κόσμο εργασίας. Κάτι ακόμα που θα ήθελα να πω είναι αυτό που λέγεται ότι η εργασιακή η κοινωνική νομοθεσία ότι δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν ξέρω τι γίνεται, μήπως είναι κάτι το καλυμμένο και θα ήθελα να πω ότι έχω εντελώς διαφορετική άποψη εγώ. Αυτό που έχει ανάγκη κανείς είναι να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διοικητικά, οικονομικά κλπ. και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και έτσι η εργασιακή νομοθεσία να ισχύσει πραγματικά για να μειωθούν τα δικαιώματα τους. Και ένα τελευταίο σημείο με διάφορες νόμους ε, ε, θα πρέπει αυτοί να εφαρμόζονται γιατί πολλές φορές επίτηδες δεν υπάρχουν και κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου επιθεώρησης για να δούμε αν όλα αυτά εφαρμόζονται ή όχι. Σε πολλές σαφείς περιπτώσεις όπως την οδηγία για τους εργαζόμενους που έχουν μετακινηθεί είτε δίθαν ανεξάρτητες εργαζόμενους. Θα πρέπει λοιπόν να τα δείξουμε αυτά στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τζιν Λάμπερτ, τους Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Υπάρχουν ένα-δυο σημεία, υπάρχουν μάλλον αρκετά σημεία από αυτά που έχουμε μπροστά μας με τα οποία θα συμφωνούσαμε σαφώς, αλλά θέλω να σχολιάσω αυτό που υπόθηκε για τους κοινωνικούς εταιρείους και τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους. Εάν τα δούμε αυτά από τη σκοπιά της απόφασης ε, για μια νομοθετική πράξη, την μεταφορά και μετά την υλοποίηση, σαφώς αυτό αφορά καθόλου την διάρκεια της διαδικασίας τους κοινωνικούς εταίρους. Θα έχουν ένα πλήρη ρόλο να διαδραματίσουν και να αναλάβουν εδώ. Επίσης, μας ενδιαφέρει πως κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν επίσης να διευκολύνουν την υλοποίηση, όπως το Ταμείο που καταπολεμά την διακριτική μεταχείριση και δίνει και εκπαιδευτικέ δυνατότητες, αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν καλύτερα τι αφορά ο νόμο και πώς εφαρμόζεται. Είδαμε και τα θέματα τη αδήλωτης εργασία. Αυτές οι πλατφόρμες μπορούν να μα βοηθήσουν να επιτύχουμε το στόχο μας. Εδώ λοιπόν μας ενδιαφέρει πώς προετοιμάζεται ο κόσμος και για την νομοθεσία την οποία θα καλυφθεί να εφαρμόσει. Και εδώ θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποια προγράμματα εκπαίδευσης, αλλά αν σκεφτούμε τις προσωρινές μορφές εργασίας, τις απροειδοποίητης εργασίας, όλες αυτές τις μορφές ε, επισφαλούς εργασίας, ε, θα πρέπει οι εργαζόμενοι και να εκπαιδευτούν για να βεβαιωθούν ότι οι νόμοι στην περίπτωση του εφαρμόζονται. Αλλά θα τα σκεφτούμε όλα αυτά και θα φροντίσουμε να υποβάλουμε γραπτώ και τι κατάλληλε τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μπεγκίν από την FTD. Δεν είναι εδώ, κανεί δεν του εκπροσωπεί. Οπότε η κυρία Μάρα Μπιτζότη. Μπιτζότο, όχι από την ΕΝΕΦ δεν θέλετε το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι τοποθετήθηκαν όλες οι πολιτικές ομάδες. Ίσως ο κύριος Κάλσον Κέμπης ε, που είναι διευθυντής τμήματάρχης εδώ να μας μιλήσει. Ευχαριστώ. Είμαι αναπληρωτής τμήματάρχης του, της Υπηρεσίας για την Εφαρμογή του Κοινωτικού Δικαίου. Σας ευχαριστούμε για την πολύ καλή σας έκθεση. Την καλωσορίζουμε και τις προτάσεις της και θα ήθελα και εγώ να θίξω κάποια από τα σημεία που ακούστηκαν στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα για την υλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας. Εδώ αντιμετωπίζουμε κάποιες δυσκολίες και προβλήματα με την καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά επαναλαμβανόμενα προβλήματα που το βλέπετε και στην έκθεσή μας, αναφέρεται. Καθυστερημένη μεταφορά. Αυτό δεν αφήνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να υποφεληθούν πλήρως από την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντιμετωπίσει και ακόμη ασχολείται με την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, προσφέροντα συνδρομή στα κρατημέλη όπου χρειάζεται. Καταρτίζοντας κάποια προγράμματα υλοποίηση εκ των προτέρων για να προσπαθήσει να, εντοπίσει θέματα, απορίες που μπορεί να προκύψουν στα κράτη-μέλη κατά τη μεταφορά. Είσαι κατοπινά στάδια και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει καθοδήγηση, εξηγήσει για το πώς μπορούν να ερμηνευτούν συγκεκριμένε διατάξεις και πώ μπορεί να μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι τα προβλήματα τη καθυστερημένη μεταφορά σύντομα θα μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα. Δεύτερο σημείο που απασχόλησε κατά μέλη του Κοινοβουλίου είναι η εκπόνηση της σωστής νομοθεσίας που να είναι εύστοχη για όλους μας, όπως και η ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των ενδιαφερομένων όλων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνοντα τη δέσμη μέτρων για την καλύτερη νομοθεσία φέτος το Μάιο, ανοίγει την ε, προοπτική, το δρόμο για την ε, ευρύτερη και καλύτερη συμμετοχή στι διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων και σε όλα τα στάδια της σύλληψη και της εκπόνησης της νομοθεσίας. Έχουν πολλές ευκαιρίες οι ενδιαφερόμενοι, τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Και η απόκριση που έχουμε από την εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας και αυτή αποτιμάται και βλέπουμε κατά πόσον η υπάρχουσα νομοθεσία εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο αρχικά ε, σχεδιάστηκε. Προσπαθούμε να περιορίσουμε το διοικητικό φόρτο, ιδίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, όπου μπορεί να εντοπιστεί αυτό, και προκύπτουν και κάποια συμπεράσματα από τις ενδεχόμενες παραβιάσεις κατά τη φάση της ε, ε, υλοποίησης και μεταφοράς, οπότε και αυτά τα αξιοποιούμε για να πετύχουμε το στόχο της καλύτερης κατανόησης της νομοθεσίας. Ευχαριστούμε στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Εάν όχι, η εισηγήτρια θέλει να προσθέσει κάτι. Παρακαλώ. Ε, przewodnicząca. Bardzo dziękuję za ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτές τις επικοδομητικές παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για όσα είπε. Αφορά την ποιότητα των κατευθυντήριων καθώς επίσης και την αποδοχή διότι η εφαρμογή τους είναι μακροπρόθεσμη ενώ ταυτόχρονα η κοινωνική εταίροι για το 2014 η Κομισιόν έκανε νέα βήματα τα οποία ε, προτάθηκαν ε, από ε, άτομα, από οργανώσεις, ε, και έτσι λοιπόν από την πλευρά της Κομισιόν καλύφθηκε σε εύρος το συγκεκριμένο θέμα. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα ε, διό, όσον αφορά τις υπάρχουσες νομοθεσίες διότι ήδη έχουμε πάρει θέση σχετικά με αυτό το θέμα Εάν λοιπόν θέλουμε να λάβουμε κάποια μέτρα σε αυτό το τομέα, τότε θα χρειαστεί ε, μία ξεκάθαρη ανάλυση των μεμονωμένων ζητημάτων. Έχω ένα σχόλια σχετικά με τα κενά στην νομοθεσία και αυτό αφορά και την ποιότητα των ε, οδηγιών. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Τώρα όσον αφορά τις αλλαγές νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό μέχρι την 8η Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν. Οπότε η 8η Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και θα υιοθετηθεί στη ε, στη συνεδρίαση της 17ης και 18ης Φεβρουαρίου του χρόνου και στη συνέχεια το Μάιο το 2016 θα συναντηθούμε, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα η Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τη συνεισφορά σας. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο αφορά την γνωμοδότηση για την εφαρμογή των συστάσεων του Κοινοβουλίου του 2010 σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική ευθύνη και θα δώσω τώρα στον λόγο ε, στην συντάκτρια της γνωμοδότησης, την Τζιάννα Μπεκίν. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο ψήφισμα 2010 για τα στάνταρτα κοινωνικά και περιβάλλοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την κοινωνική ευθύνη αυτή, οι απαντήσεις είναι σαφείς. Πώς θα μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότερο και περισσότερος χώρος για το CSR στις διάφορες συμφωνίες. Όπως το υπενθύμησε, εγώ έρχομαι από τον επιχειρηματικό κόσμο και είμαι από την ε, αρμόδια επιτροπή. Όλα αυτά τα στάνταρ και ε, αυτά τα δικαιώματα με απασχολούν ιδιαίτερα και γι' αυτό ανέλαβα με πραγματική ικανοποίηση αυτή την έκθεση και εδώ πέρα είμαι ιδιαίτερα συνδεδεμένη, έχω ιδιαίτερη σχέση με αυτή την ε, ε, ιδέα και εργάστηκα πολύ γι' αυτό και θέλησα να επιμείνω ότι στην ε, Διεθνού Οργανισμό ε, εργάστηκα προς αυτό και θα πρέπει να αποτελούν αυτά ένα κίνητρο για μια επικύρωση και δεν υπάρχει κατάλληλη πληροφόρηση, αντίθετα λανθασμένη πάνω σε αυτά και πολλές αμφιβολίες για να τα προσυπογράψουν όλα αυτά ή να τα προωθήσουν. Δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από το δάχτυλά του. Χρειάζεται αυτά τα κοινωνικά πρότυπα, τα εργασιακά, μέσω μιας κατάλληλης πολιτικής. Θα πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση να πηγαίνουν, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην όλη εμπορική στρατηγική Trade for All για μια πολιτική που να βασίζεται σε πραγματικές αξίες και να ε, προωθούνται αυτά τα δικαιώματα και νομίζω ότι το άρθρο 208 των συνθήκων προς τα εκεί πρέπει να πηγαίνουμε για τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη και για την ε, αηφόρο ανάπτυξη και για τις ε, δεύτερη συνολογή, πώς όλα αυτά επηρεάζουν. Υπάρχουν βέβαια φιλόδοξα στοιχεία, αλλά υπάρχουν και κυρώσεις, επαναλαμβάνουμε, για όσους ε, δεν τα σέβονται. Επίσης, πώς επηρεάζουν τα πράγματα για την εφόρα αυτή ανάπτυξη. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται ελέγχοι πριν και μετά τις συνθήκες, αλλά να τις συμφωνίες αλλά κυρίως πριν, ώστε να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν να υπάρξει κατάληξη. Και θεώρησα ότι από την Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσουμε μια νέα στρατηγική για την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης. Το 2010 τι ζητήσει η, το Κοινοβούλιο. Τα διάφορα κράτη να ανταποκρίνονται σε αυτά που έπρεπε, αλλά η απάντηση δεν ήταν ικανοποιητικοί, γιατί έλεγαν ότι με διάφορες άλλες χώρες ε, δεν έχουμε δεσμευτικές συμφωνίες. Πολλή εργασία που θα πρέπει να γίνει σε πάρα πολλά μέτωπα. Περιμένω τη βοήθειά σας και από τους κοιόδους ηγητές και με την ε, εισηγήτρια συνάδελφο από την ε, άλλη επιτροπή. Περιμένω τη συνεργασία της. Επίσης, τη γραμματεία ναι, ευχαριστήσω για αυτή την πολύτιμη βοήθειά της για τη σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Ε, thank you. Ε. Ευχαριστούμε κυρία Μπαγκίνη. Και τώρα ο λόγος στους σκιώδεις Αλλά δεν βλέπω εδώ την ε, συνάδελφα του ΕΛΚ, τη Σοφία Ριμπέιρο. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Συμμερίζομαι αυτά που είπε προηγουμένως η συνάδελφος, πώς τίθεται το όλο θέμα και πώς βλέπουμε αυτά τα σημεία τα οποία ειδικά μας ενδιαφέρουν και που χαράσουν πραγματικά όλη αυτή η συζήτηση στις επιτροπές του Κοινοβουλίου σχετικά με το τι θέλουμε να προωθήσουμε, τι θέλουμε να εφαρμόσουμε τι θέλουμε να συμμεριστούμε. Να προτείνω όμως κάτι. Την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών να έχουμε κάποιο χρονικό διάστημα παραπάνω και να δούμε πώς οριστικά τελικά θα μπορούσαμε να έχουμε και από την Επιτροπή Ίντα του Κοινοβουλίου να έχουμε τη σχετική γνωμοδέτηση παρόλο που η συνάδελφος είναι, συμμετέχει και στις δύο επιτροπές και αυτό στη εργασία μας να είναι ε, συνεπέστερη, ακριβέστερη επειδή είναι σημαντικά τα θέματα αυτό, αυτά και γι' αυτό λοιπόν μήπως να αναβάλουμε μετά από την παρουσίαση της ε, έκθεσης τον χρονικό όριο της υποβολής τροπολογιών μας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέρικε από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ε, προσχέδιο της ε, γνωμοδότησή σας. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι ε, εργαζόμαστε σχετικά με την κοινωνική, εταιρική κοινωνική ευθύνη εδώ μέσα και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο εδώ με αυτό το θέμα. Όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να προειδοποιήσω ότι σχετικά με το σημείο 7 ε, όλοι ε, θέλουμε να έχουμε μια ζωντανή και επιχειρηματική υπευθυνότητα, όμως ταυτόχρονα θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το, το νομοθετήσουμε. Αντιθέτως, μπορούμε να, να καταστρέψουμε με την ομοθεσία ε, καλά κίνητρα. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η κοινωνική, ε, εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να είναι εθελοντική ιδιαιτέρως όταν αφορά σε παγκόσμιο επίπεδο και σε αυτό το επίπεδο λοιπόν θα ήθελα μια περισσότερη μεγαλύτερη ανασχόλη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αναρωτηθούμε ε, τι είναι η πραγματική εταιρική κοινωνική ευθύνη και σε αυτό το σημείο λοιπόν υποστηρίζω ε, την ιδέα ενός ε, Honorable Kaufmann και είμαι των πεπιθήσεων ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε πραγματικές αξίες. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε και αυτό είναι που υποστηρίζει η δική μου παράταξη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Αβέμπερ δεν είναι εδώ. Κάποιος άλλος στη θέση της. Όχι. Ο κύριος Μέσαριτς από τους Πρασίνους δεν είναι εδώ. Η Τζιν Λάμπερτ ίσως εκ μέρους του. Παρακαλώ. Um, want... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία, κάποια σχόλια. Το, σχόλια. το ένα αφορά το πώς θα τετεριάξουμε όλα αυτά με τους στόχους ε, τη βιώσιμας ανάπτυξη που υποτίθεται είναι παγκόσμια, όχι μόνο για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ε, για ε, όλους μας και πώς αυτό αντικατοπτρίζεται σε εμάς και πώς συνδέεται με ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Όταν ε, κοιτάμε τις αξίες που αναφέρει ο συνάδελφος, νομίζω ότι όλα αυτά είναι σημαντικά, όμως ταυτόχρονα αφορά και πώς θα διασφαλίσουμε το πώς οι επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν αυτές τις αξίες δεν αντιμετωπίζονται μειονεκτικά στον επιχειρηματικό κόσμο σε αντίθεση με αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κακές πρακτικές και δεν συμμετέχουν εθελοντικά και έτσι προσπαθούν να δυσχεραίνουν την κατάσταση για τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να προωθήσουν αυτές τις αξίες. Επίσης ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και το κοινωνικό ενδιαφέρον που αυξάνεται για το συγκεκριμένο ζήτημα Κάποια από τα ερωτήματα, για παράδειγμα το εμπόριο ένδυσης, Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει μια κοινωνική γνώμη η οποία ζητά τις επιχειρήσεις ε, να τηρούν τα, ε, τα καλύτερα πρότυπα και συμφωνώ με την εισηγήτρια της γνωμοδότησης ε, που λέει ότι όλο αυτό πως ταιριάζει με την νέα ατζέντα εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα προωθήσουμε κάποιες από αυτές τις ιδέες, όχι απλά να τις ε, ε, βάλουμε ε, για ορισμένες εταιρείες και επιχειρήσεις νης που είναι ξεχωριστές στην αγορά. το πώς συνεργάζονται με τους υπαλλήλους τους και με τους συνεργάτες τους. Οπότε ανυπομονώ να το ακούσω αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε κυρία Μπερμέχιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συγχαρτήρια στην εισηγήτρια για αυτές τις προτεραιότητες που έθεσε στη γνωμοδότησή μας, στη γνωμοδότησή της, τη συμμεριζόμαστε. Να τονίσω κάτι. Την ε, συλλογική ε, εταιρική ευθύνη. Θα πρέπει να δούμε μια διπλή στρατηγική. Πώς θα ενισχύσουμε αυτά που ισχύουν ήδη και να αποκλείσουμε τις πολυεθνικές που δεν πληρώνουν, που εκμεταλλεύονται το εργαζόμενους και καταστρέφουν το περιβάλλον. Και υπάρχουν πολλές πολυεθνικές που ακολουθούν αυτές τις πρακτικές και για το σεβασμό των θεμελιώδων δικαιωμάτων. Εδώ δεν θα πρέπει να είναι απλά και μόνο ένα χνάρι, θα πρέπει να προχωράει περισσότερο και γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε η συμμετοχή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας σε αυτές τις ε, ε, διαπραγματεύσεις ε, και να είναι όλα αυτά που θα ισχύσουν δεσμευτικά. Δεν μπορούμε να είμαστε παθητικοί στα όσα θα ισχύσουν και εδώ και στην εσωτερική αγορά ή θα είτε στην εσωτερική αγορά ή θα είτε στην εξωτερική αγορά να ισχύσουν αυτά τα λανθασμένα χωρίς κάτι το δεσμευτικό, το κοινό για τις εργασιακές ακριβώς υποχρεώσεις, χωρίς τη συμμετοχή και την αναγνώριση των ε, κοινωνικών ε, των, εκπροσώπων των ε, εργαζομένων. Δεν θα υπάρχει ένα κατοθετικό στο εμπόριο. Θα πρέπει να δούμε και το τι ακριβώς απορρέει σχετικά με την αηφόρα ανάπτυξη και το πράσινο εμπόριο. Επίσης θα πρέπει να το καταφέρουμε να υπάρχουν και κοινωνικές ρήτρες και περιβάλλοντας αυτές τις συμφωνίες του εμπορίου και να είναι πραγματικά δεσμευτικές θα ε, το επαναλάβω. Και κάτι που δυστυχώς ε, γίναμε μάρτυρες, ε, ότι διατηρούμε σχέσεις σύνδεσης με κράτη τα οποία παραβιάζουν σταθερά μόνιμα διεθνώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την Δυτική Σαχάρα και για το Μαρόκο ας πούμε τα προβλήματα δεν λαμβάνονται υπόψη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ. ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση αυτή δεν μας δημιουργεί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα και στο σύνολο των παρατηρήσεων της συγκήτριας τη συμμεριζόμαστε. Thank you. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Φορμεντίνη. Όχι. Κανείς δεν είναι εδώ. Τότε θα πρέπει να σας πω απλώς το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Τζέντιλε ζήτησε μια νέα προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Όμως έχει ήδη αποφασιστεί να ισχύσει εξή προθεσμία 15 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι έχετε κερδίσει 6 μέρες παραπάνω όλοι έχουμε κερδίσει 6 μέρες έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης 25 Ιανουαρίου σχέδιο έκθεση στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 15 Φεβρουαρίου και για την Ολομέλεια δεν ξέρουμε, αλλά μάλλον θα περάσει τον Απρίλιο. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά. Να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της μερισσίας διάταξης. Δηλαδή αυτό που θα γίνει μετά το γεύμα. Σας ευχαριστώ για την πρωινή αυτή συνεδρίαση. Απλώς να σας θυμίσω ότι έχουμε προσκαλέσει πολλούς στην ακρόαση το απόγευμα που θα ξεκινήσει στις 2 κάποιες φορές άλλο χρονογρα... άλλη χρονοφυρίδα έχουμε αλλά σήμερα αρχίζουμε στις 2 το ζητήσατε εσείς το ζητήσατε από τις πολιτικές ομάδες. Ε, είναι πολύ προσκεκλημένοι μας, οπότε πραγματικά ελπίζω ότι θα έρθετε. Στις 2 το απόγευμα. Δεν είναι η συνήθις ώρα. 2. Ευχαριστώ πολύ για την συνεδρίαση ως τώρα.